ξεκινήσουμε με το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη, γιατί ο εισηγητή μα ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμο, ο κύριο Μάρκ Ταραμπέλα. Η έκθεση είναι το πρόγραμμα ενίσχυσης για τα φρούτα και τα απορροκυπευτικά όπως επίσης και τις μπανάνες και το γάλα ε, και τη διανομή του στα σχολεία. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον εισηγητή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, πράγματι είμαι έτοιμο. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, με μεγάλη περηφάνεια σα παρουσιάζω σήμερα το νέο καθεστώ ενίσχυση για την διανομή απορρεκυπευτικών φρούτων και γάλακτο στα σχολεία. Μετά από ένα χρόνο δουλειά, πρόκειται για έντονε εργασίε μεταξύ του, ε, του υποφαινομένου και των σκιωδών εισηγητών, του οποίου θα ήθελα να ευχαριστήσω. Η κυρία Ριμπέιμπορ, ο κύριο Νίκολσον, η κυρία Μίλλερ, ο κύριο Ροντρίγκε, Ρόπερ, Τζούλο και Μαρκάτη. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έκανε μια εξαιρετική πρόταση και την ε, Λουξεμβουριανή Προεδρία από τον κύριο Φρόκ Σμιτ ε, με τον οποίο συνεργαστήκαμε στενά. Σε γενικέ γραμμέ, ε, το νέο πρόγραμμα βασίζεται σε δύο πυλώνε. Ο ένα είναι η υγεία των παιδιών και η εκμάθηση υγιών συνηθιών από το σχολείο ήδη στη διατροφή του. Ε, στον πρώτο πυλώνα ε, φροντίσαμε ώστε η διανομή των οπορακεπευτικών των φρούτων και του γάλακτος να είναι υποχρεωτικά για τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Τα κράτη-μέλη συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αλλά να υπενθυμίσω ότι η συμμετοχή είναι προαιρετική. Επίση, έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν τον κατάλογο των προϊόντων, αλλά με βάση πολύ αυστηρέ προποθέσει. Παραδείγματο χάρη, απαγορεύονται οι χρωστικέ και τα τεχνητά αρώματα. Επομένως εδώ θα πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και οι εθνικές αρχές δημόσιας υγείας. Ένα από τα σημαντικά στοιχεία του προγράμματος είναι να καταπολεμήσουμε την παιδική υπαρχισαρκία και να βελτιώσουμε την υγεία των παιδιών. Τα εκπαιδευτικά αυτά μέτρα, τα οποία θα είναι υποχρεωτικά από εδώ και πέρα, θα προσεγγίσουν και τα παιδιά στη γεωργία, μαθαίνοντα ε, επίση και καλές συνήθειες από παιδιά. Ε, μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξουν ε, ε, συνήθειε υγιή τα παιδιά και επομένω θέλουμε να βοηθήσουμε επίση και την τοπική και την περιφερειακή παραγωγή, τα βιολογικά προϊόντα και να βοηθήσουμε του τοπικού παραγωγού και να δίνονται προϊόντα με βάση την εποχικότητά τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Το Συμβούλιο ήθελε να εφαρμοστεί το άρθρο 43.3 και να μας αποκλείσει από αυτό το θέμα, αλλά τελικά στις διαπραγματεύσεις ε, είχαμε τη βάση 43.2 που περιλαμβάνει συναπόφαση με τη βοήθεια όλων των σκιωδών εισηγητών καταφέραμε να ε, προασπίσουμε τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου. Και στον προπολογισμό έχουμε αύξηση του θέματος αυτού κατά 20 εκατομμύρια ευρώ για ε, το γάλα γιατί υπάρχουν χώρες που χρησιμοποιούν ε, το πρόγραμμα εδώ και καιρό και δεν θα πρέπει να τιμωρωθούν επειδή ε, θα δοθεί η δυνατότητα αυτή σε χώρες που δεν έχουν ιστορική ε, χρήση γάλακτος στα σχολεία, όπως για παράδειγμα η Κροατία που θα ενταχθεί τώρα. Προσπαθούμε να δούμε και τι γίνεται. Έχει δοθεί ένα 5% επιπλέον για τις υπερπόντιες περιοχές. Κάποιοι ήθελαν 40%. 40% δεν έχει νόημα. Δεν θα σταματήσει ένα πρόγραμμα εις βάρος κάποιου άλλου ή προ όφελο κάποιου άλλου. Επομένω, ε, καταφέραμε να υπάρχει συγκεκριμένη ε, διανομή ε, βάσει και τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να γίνει κατάλληλη κατανομή του προπολογισμού μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχουν δύο κριτήρια για όλο το πρόγραμμα. Να δίνονται σε παιδιά 6 έως 10 ετών στα κράτη-μέλη και επίσης να υπάρχουν και μέτρα αναπτυξιακά στις διάφορες περιφέρειες των κρατών μελών. Ε, όπως σας είπα, είναι ιστορικές ε, βέβαια και οι πτυχές που εφαρμόζονται. Δεν θα πρέπει βέβαια να ξεχνάμε και χώρες που δεν έχουν ιστορικές αναφορές. Ε, θα πρέπει να λαμβάνουμε και αυτές υπόψη. Η προβολή των προγραμμάτων και η ε, μείωση του γραφειοκρατικού έκθους είναι προτεραιότητα για το Κοινοβούλιο, ώστε να έχουμε όλο και μεγαλύτερο αριθμό σχολείων και παιδιών που θα αποφελούνται από το πρόγραμμα. Γι' αυτό ακριβώ ζητώ από του συναδέλφου να υποστηρίξουν την έκθεση αυτή που θέλει να βελτιώσει την υγεία των παιδιών, να του ε, μάθει νέα πράγματα για την υγεία και τη διατροφή του και φυσικά να βοηθήσουμε τον τομέα των απορροκυπευτικών και των φρούτων. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ταραμπέλα. Ο λόγος στον Επιτροπό Χόγκαν, εκ Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ όλους και ιδιαίτερα τον κύριο Ταραμπέλα και τους σκιώδεις ηγητές για την εργασία τους. Είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Ταραμπέλα και οι σκιώδεις ηγητές θα συμφωνήσουν ότι αυτή ήταν μια πολύ περίπλοκη διαδικασία έπρεπε να λυθούν σημαντικά θέματα όπως τα, ποια προϊόντα θα καλύπτονται, το χρονοδιάγραμμα, οι μεταφορές ε, και η νομική βάση. Μετά από μακροσκελή συζήτηση, νομίζω ότι εξασφαλίσαμε μια ισορροπημένη συμφωνία. Χάρη σε μεγάλο βαθμό τη συνεισφορά του Κοινοβουλίου. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί μόνο μέσω ε, ευελιξία από όλες τις πλευρές και επικοδομητική τάση. Εμείς ε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να συνεχίσουμε την ε, διαδικασία αυτή στο μέλλον. Ε, νομίζω ότι το Κοινοβούλιο βοήθησε στο να ενισχύσουμε το θέμα της ασφάλειας. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στα νοπά προϊόντα. Επίσης, για τους στόχους, στο, ένας από τους στόχους είναι ότι τα παιδιά θα πρέπει να μάθουν να αξιολογούν και να εκτιμούν την αξία αυτών των προϊόντων. Ελπίζω ότι αύριο θα επιβεβαιωθεί στην ψηφοφορία η επένδυση 250 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως ε, για την, ε, σε μια περίοδο 6 ετών λοιπόν θα έχουμε πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα αυτό γίνεται σε μια περίοδο πολύ δύσκολη για τους μας, μας, ιδιαίτερα στον τομέα των γαλακτοκομικών. Η αύξηση αυτή θα δώσει βοήθεια και στον τομέα και θα ε, βοηθήσει τα παιδιά να δημιουργήσουν υγιείς, συνθήκες, ε, να πάρουν υγιείς ε, συνήθειες για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. έχει το λόγο καταρχήν. Για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ όλους που συνέβαλαν στο να έχουμε ένα βελτιωμένο πρόγραμμα διανομής γάλακτος και επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω προσωπικά τον εισηγητή και τους σκιώδη εισηγητές. Σε πέντε τριμερείς ε, τριγωνικές συζητήσεις ε, καταλήξαμε μετά από πέντε, καταλήξανε όλοι ότι συμφωνούν μαζί μου. Άρα δηλαδή αυτό που τίθεται τώρα επιτάπητος είναι να εφαρμοστούν ταχύτατα τα προγράμματα στα κράτη-μέλη. Η ε, σημασία του προγράμματος είναι ότι θα πρέπει να ενοποιηθούν τα προγράμματα και τώρα πλέον θα πρέπει να ε, μεταφερθούν κάποια σημεία προγραμμάτων σε άλλα. Αυτό το βρίσκω πολύ θετικό. Και αυτό που είναι ιδιαίτερα ευτυχές ε, είναι ότι το Κοινοβούλιο ε, αύξησε κατά άλλα 10 ευρώ και πλέον διατίθεται για το σχολικό πρόγραμμα διατίθεται 150 ευρώ. Το είπε ο κύριος ε, Ταραντέλα ότι αυτό σημαίνει ότι τα κονδύλια που εκταμιεύονται στα κράτη-μέλη παραμένουν στο ίδιο ύψο και λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η κατάσταση στην Κροατία και στις ε, εξόχως απομακρυσμένες ε, περιοχές. Θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι τα παιδιά μας ε, και τα σχολεία μας συμμετέχουν πλέον στα θαυμάσια προϊόντα μας και προβλέπεται επίση κάποια κονδύλια να διατίθενται για λόγους εκπαιδευτικούς. Και αυτό είναι απολύτως απαραίτητο έτσι ώστε να μάθουν τα παιδιά ότι το γάλα δεν έρχεται από την ε, μόβα γελαδίτσα που απεικονίζεται στις σοκολάτες αλλά από μια πραγματική αγελάδα που βόσκει στα χωράφια, τα λιβάδια. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντεκάστρο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, το πρόγραμμα διανομής ε, φρούτων και γάλακτος στα σχολεία είναι ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενθαρρύνονται τα παιδιά να έχουν υγιεινή διατροφή και να καταναλώνουν τα παραδοσιακά προϊόντα μας. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον κύριο Ταραμπέλα και όλη τη διαπραγματευτική ομάδα για την θαυμάσια δουλειά που έκαναν και για το εξαίσιο αποτέλεσμα που πέτυχαν. Πέτυχαν για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον σημαντικό δημοκρατικό του ρόλο ως συνομοθέτης και επ' αυτού επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω και την Επιτροπή η οποία τήρησε και σεβάστηκε θέση του Κοινοβουλίου μέχρι τέλους. Παρ' όλα αυτά βέβαια η επιλογή του Κοινοβουλίου να τεθούν σε συζήτηση σημαντικά σημεία της αρχικής πρότασης αυτό οδηγεί στο να υπάρχει ένα επίμαχο, ε, μια επίμαχη συμφωνία που δεν ξέρω κατά πόσο θα καταλήξει πράγματα ώστε να υπάρχει πιο ίση και αναλογική κατανομή του, των προϊόντων στα κράτη-μέλη. Αυτό που ενδιαφέρει όμως είναι η διατροφική, ο διατροφικός πολιτισμός ε, να είναι ένα σημαντικό κομβικό στοιχείο που θα αφορά στην εκπαίδευση των νέων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Νίκολσον για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να, εισηγη... να συγχαρώ τον εισηγητή για την πάρα πολύ καλή δουλειά. Υπάρχουν δύο μικρό προβληματάκια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας ε, ξέσιος ε, εισηγητής, αλλά και όλοι οι άλλοι που συνεργάστηκαν μαζί του. Εγώ χαιρετίζω την πρόταση. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή, είναι ισχυρή, εκπέμπει ισχυρά μηνύματα, όχι μόνο στο γαλακτοκομικό τομέα, αλλά και στον τομέα των φρούτων. Οι αποφάσει που λήθησαν είναι το Κοινοβούλιο συνέβαλε τα και αυτό αποδεικνύει ότι οποτεδήποτε υπάρχει συνεργασία είναι δυνατόν να επιτευχθούν πολλά περισσότερα από αυτά που πίστευε κανείς αρχικά. Εν πάση περιπτώσει εγώ προσβλέπω στην εφαρμογή του προγράμματος γνωρίζω ότι τα περισσότερα μέλη της ομάδας ECR ε θα υπερψηφίσουν η πρότασή σας θα περάσει και επίσης επιτρέψτε μου να πω ότι όσον αφορά το θέμα του προπολογισμού αυξήθηκαν τα κονδύλια ε, και βέβαια να πω και κάτι σήμερα το βράδυ χαίρομαι που έχουμε αυτή τη συζήτηση αλλά είναι λυπηρό το ότι δεν θα έχουμε τη συζήτηση για τα γουρούνια, για τους χείρους ε, το κοινοβούλιο αυτό ε, θα έπρεπε να κάνει τη συζήτηση ενώπιον του Επιτρόπου δεν νομίζω ότι αυτό βέβαια θα σήμαινε ότι δείχνουμε έλλειψη σεβασμού στον εισηγητή ο οποίος έτσι και έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά ο κύριος Κύριε Νίκολσον, έχουμε ένα συνάδελφο ε, που ε, θέλει να σας υποβάλει μια ερώτηση. Δέχεστε, Τζιμ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που δέχεστε την ερώτησή μου, κύριε Νίκολσον. Δεν είστε εσείς, λοιπόν, κύριε Φροντζελίκα. Την επόμενη φορά εσείς. Συνάδελφε. Ναι, πολύ σημαντικό εκπαιδευτικά το πρόγραμμα αυτό για τα παιδιά, συμφωνώ. Όμως ο τίτλος αυτής της έκθεσης που δίνει έμφαση στις μπανάνες, δηλαδή μιλάμε για απορροκυπευτικά και γάλα, αλλά βάζουμε και τις μπανάνες. Δεν θα έπρεπε να δίνουμε πιο πολύ έμφαση στα μήλα για παράδειγμα, που είναι ευρωπαϊκή παραγωγή. Να πούμε, απορροκυπευτικά μήλα, μπανάνες και γάλα. Δεν θα πρέπει να στηρίξουμε την ε, ευρωπαϊκή παραγωγή. Κύριος Νίκολσον. Ε, ευχαριστώ για αυτήν την εξαιρετική ερώτηση. Δεν θα είχα πρόβλημα να βάλουμε όλα τα φρούτα, να τα παριθμίσουμε και τα αχλάδια και τις φράουλες και ό,τι θέλετε. Οπότε δεν θα είχα πρόβλημα. Εμείς, εγώ έρχομαι από το Κάρντιφ στην Βόρεια Ιρλανδία. Εκεί πράγματι παράγουμε πάρα πολλά μήλα. Είμαστε η πατρίδα του μήλου. Οπότε <laughs> με πολύ χαρά θα δεχόμουν την πρόταση αυτή. Ε, ευγενές φρούτο. Um, Ευχαριστώ. Δύο λεπτά κυρία Μίλλερ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Ταραμπέλα για την ε, πάρα πολύ καλή δουλειά που έκανε στο πλαίσιο των τριμερών συζητήσεων. Ε, πραγματικά μπόρεσε, κατόρθωσε να διατηρηθούν οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ βέβαια και τους και ηγητές. Κατορθώσαμε να διατηρήσουμε και να εγκρίνουμε τον κανονισμό για τα φρούτα και το γάλα στα σχολεία. Ελπίζω να υπάρξει μεγάλη πλειοψηφία υπέρ αυτής της πρότασης. Ε, πρέπει να κατορθώσουμε να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία. Επιτύχαμε την αύξηση των κονδυλίων και αυτό δεν ήταν προφανές ε, στην αρχή. Με αυτό λοιπόν το πρόγραμμα ε, θα έχουμε πρόσβαση σε 30 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών τα οποία ε, κάθε εβδομάδα ε, θα παίρνουν δωρεάν γάλα και φρούτα. Για μένα δύο πράγματα είναι σημαντικά. Το ένα είναι να συμπεριληφθεί και ο κατάλογος των μεταποιημένων προϊόντων και το δεύτερο είναι τα συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα σχετικά με τον διατροφικό πολιτισμό. Στο μέλλον ε, θα μπορούσε να πηγαίνουν διατροφολόγοι στα σχολεία για να μεταφέρουν ε, τις γνώσεις τους στα παιδιά. Γιατί από ό,τι φαίνεται έχουν γίνει κάποια λάθη τα παιδιά μας ε, κάπως δεν ελέγχουν την καθημερινότητά τους, δεν γνωρίζουν πώς χειρίζεται κανείς τα βασικά ε, διατροφικά προϊόντα και πώς με αυτά μπορεί κανείς επίσης ε, να ετοιμάσει το καθημερινό φαγητό. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο κατορθώσαμε να το εμπεδώσουμε στα προγράμματά μας και χαίρομαι πάρα πολύ που τα συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα θα οδηγήσουν στην ε, καλή κατάσταση και στην καλή υγεία των παιδιών. Εμείς ε, δεχόμαστε το αποτέλεσμα του τριγωνικού διαλόγου με πολύ μεγάλη χαρά. Κυρία Μίλο, έχουμε μία μπλε κάρτα από την κυρία Γκραπίνη. Τη δέχεστε, μάλιστα. Κοιτάξτε, και εγώ συμφωνώ πάρα πολύ ότι η υγεία των παιδιών είναι προτεραιότητα και συγχαίρω τον κύριο Ταραμπέλα, αλλά θέλω να υποβάλω μία ερώτηση που έχει σχέση με το να προσφέρουμε μεγαλύτερη υποστήριξη στα παιδιά ηλικία 6 και 10 ετών. Και πώ καταλήξατε στο 6 μέχρι 10 και δεν είπατε 10 με 14. Εγώ νομίζω ότι το ηλικιακό φάσμα θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερο. Αγαπητοί συνάδελφε, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Κοιτάξτε, γενικά βεβαίως και όλοι μας ε, είμαστε υπέρ του να μπορούν όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα τρόφιμα. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι τα παιδιά που είναι στις πρώτες τάξεις του σχολείου. Σε τελική ανάλυση όλα εξαρτώνται από τα χρήματα. 1,5 δι σε 6 χρόνια εκταμιεύτηκαν, νομίζω ότι είναι ικανοποιητικό το ποσό ε, και τα κράτη-μέλη αν θέλουν μπορούν γιατί όχι να συγχρηματοδοτήσουν. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Σένερα Ροντρίγκεφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ταραμπέλα για τη δουλειά του. Ε, εκτιμούμε θετικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να υποστηρίζει την διανομή φρούτων ε, μπανάνας οποροκυπευτικών και γαλακτοκομικών στο σχολείο ως τρόπο να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά για το ρόλο των οπών προϊόντων στην διατροφή και να μάθουν και την προέλευση των προϊόντων. Ήταν πολύ θετικό το γεγονός ότι έχουν συμπεριληφθεί και η δυνατότητα να δυθούν κίνητρα για τοπικά προϊόντα και βιολογικά προϊόντα. Για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση με τον τρόπο, για τον τρόπο με τον οποίο έχουν παραχθεί αυτά τα προϊόντα και πώς βοηθούν την οικονομία και πώς μπορούν μπορούν να βοηθήσουν ε, να διατηρηθεί ε, ζωντανή η αγροτική παραγωγή. Επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε και επισκέψεις σε γεωργούς, άνδρες και γυναίκες και στις τοπικές αγορές ε, για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε και το σημείο, άρθρο, το σημείο 2.9 αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ για δυόμιση λεπτά ο κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε, κυρίε και κύριοι, να ευχαριστήσω τον κύριο Ταραβέλα καταρχήν. Πολύ καλή δουλειά του. Ήμουν σκιώδης εισηγητή εκ μέρους των Πρασίνων. Παρόλο ότι αρχικά δεν ταυτιζόμουν με τον εισηγητή πλήρως, το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Γιατί και γιατί αξίζει να το υποστηρίξουμε. Να πω καταρχήν ότι καθορίζει στόχους ε, για την ανάπτυξη καλών συνηθιών. Επίσης διευρύναμε τον κατάλογο των προϊόντων που θα χορηγούνται και αυτό έχει σχέση και με την ενημέρωση των μαθητών και με τις υγιεινές συνθήκες. Τώρα, ίσως είναι υπερβολικά ευρύς ο κατάλογος βέβαια. Πώς είναι να τον κανείς να φάει ελαιόλαδο ε, και ποιες είναι οι καλές, συνθήκες, ε, οι καλές συνήθειες που ε, δίνουμε στα παιδιά όταν τους επιτρέπουν να πίνουν γάλα με σοκολάτα. τέλο πάντων. Για πρώτη φορά σε μια νομική πράξη αναφέρεται ότι το μονοσόδιο, η γλουταμάτι μονοσόδιο ε, και άλλους τέτοιους, τέτοιες βελτιωτικές ουσίες δεν θα πρέπει να, να χρησιμοποιούνται. Έτσι κι αλλιώς ε, δεν θα ήταν λογικό, φαίνεται αυτονόητο, αλλά δεν ήταν τόσο απλό. Επίσης βελτιώσαμε τη συνολική διαχείριση του έργου αυτού. Στο καινούριο έγγραφο έχουμε διευκρινίσει τα κριτήρια για, την, ε, για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιούνται τα ποσά της χρηματοδότησης και επίσης πολύ σημαντικό για τη διαχείριση οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές θα έχουν μεγαλύτερη εμπλοκή τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή των μέτρων. Και αυτό είναι σημαντικό διότι οι τοπικές αρχές συνήθως γνωρίζουν πολύ καλύτερα τις τοπικές ανάγκες. Ευχαριστώ. Ο ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον συγγητή τον κύριο Ταραμπέλα για την εξαιρετική του δουλειά και για τον τρόπο με τον οποίο διεξήγαγε για τις διαπραγματεύσεις στον τριμερή διάλογο. Διαπραγματεύσεις οι οποίες επέτρεψαν να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα κατά την άποψή μας. Καταρχάς όσον αφορά τον προπολογισμό, επομένως το κατάλληλο ποσό για το πρόγραμμα διανομής ε, οποροκυπευτικών φρούτων και γάλακτος στα σχολεία, αλλά επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικός ο στόχος. Ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει. Να εκπαιδεύσει τα παιδιά να καταναλώνουν νοπά προϊόντα, περιορίζοντας τη χρήση σακχάρων και πρόσθετων αλάτων. Διότι σε μία ήπειρο όπου το 26% των ενηλίκων είναι παχύσαρκο, ε, είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε από τα σχολεία. Να ξεκινήσουμε από τα σχολεία ώστε να διδάξουμε και να κατανοήσουν τα παιδιά πώ μπορούν να έχουν μια υγιεινή, υπεύθυνη και βιώσιμη διατροφή. Όταν θα πρέπει να εφαρμοστεί το πρόγραμμα δεν θα πρέπει να σταματήσουμε. Φυσικά θα πρέπει να βεβαιωθούμε στα κράτη-μέλη ότι θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα με τον καλύτερο και ορθότερο δυνατό τρόπο και θα γίνουν όλοι απαραίτητοι έλεγχοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Τζούλο, υπάρχει ερώτηση από τον ε, ε, κύριο Κουλαή. Ε, δέχεστε την ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ακούσαμε πολύ προσεκτικά τον κύριο Ταραμπέλα και άλλους να λένε ότι ο στόχος αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός, είναι καλός για την υγεία των παιδιών μας, είναι καλός για τη βιομηχανία και τη γεωργία. Ε, τα ακούσαμε όλα αυτά. Η ερώτησή μου προς εσάς είναι κατά πόσον συμφωνείτε μαζί μου ότι είναι καθήκον και υποχρέωσή μας ε, ώστε το πρόγραμμα αυτό να παρουσιάζεται ως ένα κοινό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως είναι καλό για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί μου φαίνεται πολύ περίεργο το γεγονός ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που συνεχώς επισημαίνουν τα αρνητικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναφερθούνται σε κάτι θετικό όπως αυτό. Κύριε Τσούλο, 30 δευτερόλεπτα. Δεν κατάλαβα ε, ε, ποια ακριβώς ήταν η ερώτησή σας, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ ουσιαστικό να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά, ε, ώστε οι νέοι σήμερα που θα είναι και οι ενήλικες ε, στο μέλλον να φτάσουν στην αγορά εργασίας ε, και στον κόσμο της εργασίας πλήρως συνειδητοποιημένοι. Και αυτό φυσικά νομίζω ότι είναι ένα κοινό σημείο και δεν υπάρχει διαφοροποίηση εδώ. Ο κύριος Φεράν για ένα λεπτό. Χαίρομαι που βλέπω πως η δουλειά που κάνουμε εδώ στο Κοινοβούλιο είναι πολύ συχνά καλύτερη ποιότητα από τη δουλειά που κάνει η Κομισιόν και μας προτείνει. Να πω το εξή, η συνέχιση του προγράμματος διανομής προκυπευτικών γαλακτοκομικών προϊόντων και εμπανανών στα σχολεία είναι κάτι πολύ καλό, πραγματικά πολύ καλή εξέλιξη. Όμως, Υπάρχουν ακόμα σημαντικέ δυσκολίε που αντιμετωπίζουμε. Το κείμενο αυτό επιτρέπει στα κράτη-μέλη ε, να εφαρμόσουν το πρόγραμμα όπως επιθυμούν και να ευνοήσουν τα τοπικά προϊόντα. Καλούμε λοιπόν ε, τα μέλη να στηρίξουν αυτό το πρόγραμμα και την έκθεση και ε, να ευνοήσουν την προώθηση τοπικών προϊόντων, προϊόντων από τις κοντινές κοινωνίες και ευρωπαϊκών προϊόντων. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό, λεπτό λόγο στην κυρία Ρανθ Καρθία. Αυτή η, η έκθεση που συζητάμε σήμερα είναι πολύ καλή, ωφέλιμη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα κράτη-μέλη και για το γεωργικό και κτηνοτροφικό ε, τομέα, αλλά κυρίως για τα παιδιά που θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν την γαστρονομική τους κουλτούρα και τη διατροφική τους κουλτούρα. Το γεγονός ότι ελήφθησαν υπόψη τα πολύ μικρά παιδιά επίσης είναι πολύ σημαντικό. Τα 20 εκατομμύρια που δίνουμε παραπάνω για τον, το γάλα είναι επίση πολύ θετικό. Θα πρέπει να διευρύνουμε προφανώ τον προπολογισμό εφόσον διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή. Και μετά η μεταφορά μεταξύ ε, προκυπευτικών και γάλακτος, ε, η δυνατότητα αυτή είναι πράγματι δυνατότητα στα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν τον προπολογισμό τους στην εθνική τους πραγματικότητα. Ε, καλωσορίζω λοιπόν όλα αυτά τα σημεία. Επίσης την εισαγωγή φρούτων, μεταποιημένων φρούτων διότι έτσι τα φρούτα και άλλα προϊόντα ε, γίνονται πιο εύληπτα από τα παιδιά νοπά αλλά και ε, μεταποιημένα, όπως για παράδειγμα γιαούρτι. Αργότερα η εισαγωγή ε, του ελαιολάδου, του μελιού και των ε, ελιών ε, θα μπορούσε να προσθεθεί στο μέλλον παρόλο που δεν τα καταφέραμε αυτή τη φορά. Ευχαριστώ. Έχουμε μια μπλε κάρτα για σας νομίζω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω κάτι για τον περιορισμό της ε, γραφειοκρατίας. Ε, ε, υπάρχει αυτό που λέγεται στην βίβλο πίστευε και μία ερεύνα. Όμως, ε, κρίνεται ότι μπορούν τα κράτη-μέλη να εξαναγκαστούν το πρόγραμμα αυτό να το εφαρμόζουν χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς ε, λάβαμε μία απόφαση, τώρα πρέπει να το εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη, αλλά εγώ έχω τις αμφιβολίες μου. Δεν ξέρω αν ισχύει, το πίστευε και μία ερεύνα. Querido το σημαντικό είναι τα κράτη-μέλη να ενθαρρυνθούν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα που αυτή τη στιγμή δεν είναι υποχρεωτικό. Θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό. Θα έπρεπε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια και να κάνουν την προσπάθεια τα κράτη-μέλη ώστε τα νέα και τα παιδιά να βελτιώσουν τις διατροφικές τους συνήθειες. Η γραφειοκρατία είναι ένα μόνιμο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να βρούμε μια μέση λύση ανάμεσα στην ε, ορθή ε, διαχείριση των, του προπολογισμού και στην ευελιξία. Κύριε Νόχιλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνώ και εγώ με αυτά τα οποία ελέγχθησαν. Επιτύχαμε τρία σημαντικά θέματα, δηλαδή τα προγράμματα τα οποία εφαρμόζονται επιτυχώς εδώ και πολλά χρόνια. Αυτά ενοποιήθηκαν, αυξήθηκαν επίσης τα κονδύλια, βελτιώθηκε και η νομική βάση και επιβεβαιώθηκαν οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου. Αυτό που θέλω να πω σήμερα είναι το εξή. Πρέπει να προβάλλουμε καλύτερα το στόχο. Ο στόχο των προγραμμάτων είναι σαφή ότι θα πρέπει να μάθει κανείς και με την αφή του. Στο σχολείο ε, πολλά μαθαίνονται μέσα από τις πολιστές και άλλα, αλλά ε, πρέπει κανείς ε, και τα παιδιά δηλαδή να μάθουν με τα χέρια τους, με την ε, αυτή όπως σας είπα και με τη γεύση η γεύση είναι κάτι που και αυτό παίζει ρόλο ε, τώρα πια έχουμε μόνο τα ταχυφαγεία και τα παιδιά τρώνε μόνο αλμυρά ε, δεν είναι πια σε θέση να διαφοροποιήσουν λιγάκι τη γεύση η γεύση λοιπόν είναι σημαντικός στόχος και στη τελική ανάλυση είναι σημαντικό και η αλλαγή συμπεριφοράς τα παιδιά τα οποία θα παίρνουν στο σχολείο φρούτα και γάλα αυτοί είναι οι μελλοντικοί μας καταναλωτές αυτά τα παιδιά παιδιά από την αρχή να εξοικειωθούν με ποιοτικά προϊόντα και αργότερα όταν θα είναι ενήλικες θα τα αγοράζουν. Ο κύριος Κούσνικ. Ευχαριστώ πολύ κύριε πίτροπε και εγώ θέλω να πω κάτι σχετικά με το γάλα και το πρόγραμμα για γάλα και φρούτα στα σχολεία. Πιστεύω ότι βεβαίως και είναι σημαντικό να επηρεαστούν οι συνήθειες ε, διατροφής είναι το πρώτο πρόγραμμα Μάλλον εφαρμόστηκε ήδη ένα πρόγραμμα, τώρα έχουμε ένα δεύτερο μικρότερης διάρκειας, αλλά πάντως είναι σημαντικό το ότι θα υπάρξει πρόσβαση σε πάρα πολλά σχολεία. Μήπως μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο αργά, λέει πρόεδρος. Λοιπόν, ε, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα δημοσιονομικό πλαίσιο και το Κοινοβούλιο πρέπει να προσφέρει την υποστήριξή του έτσι ώστε στο πρόγραμμα αυτό να συμμετέχουν όσο δυνατόν περισσότεροι. Γιατί είναι σημαντικό να υποφεληθούν όσο πιο πολλά παιδιά γίνεται και νέοι βέβαια έφηβοι γιατί αυτοί στο μέλλον θα είναι οι αγοραστές γάλακτος και φρούτων και κυπευτικών. Αυτοί θα είναι οι καταναλωτές μας του μέλλοντος. Τώρα θα έχουμε ε, άλλα 20 εκατομμύρια ευρώ για αυτό το πρόγραμμα ε, γάλακτος ε, στα σχολεία και 150 εκατομμύρια επιπλέον για το πρόγραμμα φρούτων και γάλακτος. Για ένα λεπτό ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι εδώ ε, έχουμε πέσει σε ένα ε, παράπτωμα παράληψης γιατί κανονικά αυτό θα έπρεπε να είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών ενώ εμείς το περνάμε για λόγους υγείας ως ευρωπαϊκό. Είμαι λίγο σκηνικό, αλλά νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να παρισφρήσει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Επίσης με ενδιαφέρον διαπιστώνω ότι τα σχολεία ε, που εντάσσονται στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ε, σε, θα παίρνουν ένα κόκκινο βραβείο ευγνωμοσύνης. Τα παιδιά πρέπει να μας λένε πόσο χαίρονται. Όσο περνάνε προς το σχολείο θα βλέπουν ε, ε λιβάδια ευγνωμοσύνης και μετά φτάνοντα στο σχολείο θα του δίνουμε και άλλα πράγματα και όλα αυτά τα πράγματα θα γίνονται στη διάρκεια του δημοψηφίσματος για την Ελλάδα. Και ελπίζω λοιπόν θα ότι θα είναι βρετανικό γάλα αυτό το οποίο θα διανέμεται και επομένως ε, τα προϊόντα του ε, θα αναφέρονται και δεν θα αναφέρονται οι μπανάνες. Κύριε Άγνιου, υπάρχει μια μπλε κάρτα για σας από τον κύριο Γιάκοβιτς. Τη δέχεστε, παρακαλώ. Μπορείτε να θέσετε την ερώτησή σας. Ευχαριστώ πολύ που δέχεστε την μπλε κάρτα μου. Είπατε ότι η υγεία θα πρέπει να είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών ε, στο εθνικό πλαίσιο, αλλά ε, σας ρωτάω πώς μπορείτε να το λέτε αυτό όταν ξέρετε τι επιδημίες αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, τη στιγμή στον κόσμο. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας μας προειδοποιεί για αυτά. Μην κατηγορείτε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η υγεία όταν υπάρχουν επιδημίες και πανδημίες ε, στην Ιφίλιο. Συμφωνείτε. Ε, ε, λέτε κατηγορηματικά ότι η υγεία είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα κράτη-μέλη είναι κάτι πολύ απλό. Είναι το μόνο από τα λίγα πράγματα που δεν ισχύουν και θα, ήθελα σε καμία περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Η κυρία Πέτυρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή. Οι διαπραγματεύσεις έλξαν ε, πολύ με μεγάλη επιτυχία. Το κείμενο αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ιδιαίτερα για τα παιδιά στην Κροατία. Το κείμενο, το τελικό κείμενο ήρε τα, τα οποία ε, δεν επέτρεπαν στην Κροατία να χρησιμοποιήσει κοινωνική χρηματοδότηση για την διανομή ε, τέτοιων προϊόντων στα σχολεία. Ε, χαίρομαι που τα επιχείρηματά μου λήθησαν υπόψη. Ε, η διαπραγματεύση αυτή θα επιτρέψει στους παραγωγούς να μπουν σε μια καινούργια αγορά με τη διανομή τέτοιων προϊόντων στα σχολεία. Επίσης επιτρέπει στα κράτη-μέλη το κείμενο να συμπεριλάβουν ένα πιο ευρύ ε, φάσμα προϊόντων ε, μεταξύ αυτών τοπικά προϊόντα όπως το λάδι, οι ελιές, το μέλι. Το πρόγραμμα αυτό δεν είναι άλλωστε μόνο εκπαιδευτικό, εκπαιδευτικό έχει και μια κοινωνική διάσταση. Γιατί για τα φτωχά παιδιά ίσως αυτό το γεύμα να είναι το μοναδικό γεύμα της μέρας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μπλε κάρτα από τον κύριο Τσάνι. Τη δέχεστε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ που δέχεστε την μπλε κάρτα μου. Να ε, ρωτήσω τη συναδελφή αλλά και τους άλλους συναδέλφους. Πιστεύω ότι σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υπάρχουν ειδικά προϊόντα, ειδικά τοπικά προϊόντα που είναι, έχουν ιδιαίτερη σημασία ε, για την κάθε χώρα. Όμως στην πραγματικότητα μιλάμε για 4 ευρώ για κάθε παιδί κατέτος. Έτσι, τόσα θα είναι τα χρήματα που θα βγαίνουν από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό για κάθε παιδί κάθε χρόνο. Δεν νομίζω ότι είναι σημαντικό ποσό αυτό, οπότε είναι λίγο σχετικά όλα αυτά. Ε, όσα, και να έχω, λεφτά και να δίνουμε, αν είναι για τα παιδιά και την ευημερία τους, ε, ευπρόσδεκτα. 250 εκατομμύρια το χρόνο ε, για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το ποσό, ε, είναι το κονδύλι. Ε, εντάξει, ασφαλώ και δεν είναι απόλυτα αρκετό. Στην Κροατία έχουμε 17.000 παιδιά τα οποία πεινάνε. Δεν μπορούν να αγοράσουν γεύματα στο σχολείο γιατί οι γονείς δεν έχουν αρκετά χρήματα. Οπότε έστω και ένα γεύμα δύο φορές τη βδομάδα θα είναι δωρεάν, οπότε θα τα βοηθήσει. Ευχαριστώ πολύ. 1,5 λεπτό στην κυρία Κάτεμπαχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ταραμπέλα και όλους τους άλλους που διαπραγματεύτηκαν γιατί νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ ικανοποιητικό. Ακούω την κριτική ότι 250 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι μεγάλο το ποσό. Ε, κοιτάξτε, κάτι είναι και αυτό και είναι σημαντικό ότι έγινε ένα βήμα προς τα εμπρός. Δηλαδή ε, χρήματα προς όφελος των ανθρώπων και των παιδιών. Τα 5 δις για τα επόμενα 6 χρόνια δεν θα είναι βοήθεια μόνο για τη γεωργία και για τα προϊόντα που παράγονται στην Ευρώπη, αλλά κατά κύριο λόγο κάτι που θα βοηθήσει τα παιδιά μας να τρέφονται υγιεινά, να δουν πόσο γευστικά είναι αυτά τα ποιοτικά προϊόντα, να απορρίψουν τα μεταποιημένα. Όλα αυτά μπορούμε να τα επιτύχουμε με το πρόγραμμά μας. Και ε, παρότι εγώ δεν συμφωνώ 100% με το συμβιβασμό, γιατί πιστεύω ότι το σοκολατούχο γάλα δεν έπρεπε να ενταχθεί, δεν συμφωνώ. Ε, εγώ θεωρώ ότι μόνο το γάλα πρέπει να προάγεται και όπως είπαν και οι συνάδελφοι ε, στο μέλλον δεν θα πρέπει να έχουμε αρωματικές ουσίες, ε, συνθετικές ουσίες αυτά τα προϊόντα. Αυτά είναι πολύ σημαντικά βήμα και να πω στο συνάδελφο Ένιου Κοιτάξτε, μάλλον δεν έχετε διαβάσει καλά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Το άρθρο 68 αναφέρεται ότι η υγεία ε, είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, άρα δηλαδή είναι σημαντικό σε όλες τις πολιτικές να λαμβάνονται υπόψη θέματα υγείας. Και ακριβώς αυτό κάνουμε εδώ, στη γεωργία, στην ε, παιδεία, στον τομέα της υγείας. Αυτά πράττουμε. Κυρία Κάρεμπαχ, ε, είναι μια μπλε κάρτα από την κυρία Μάλατιτς. Δέχεστε παρακαλώ για 30 δευτερόλεπτα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφό μας. Άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά που είπατε και συμφωνώ μαζί σας ότι αυτό το πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό για να προάγουμε τα υγιεινά προϊόντα ε, για τα παιδιά στα σχολεία και για εκπαιδευτικούς λόγους. Ερωτώ όμως, πιστεύετε ότι αυτό το πρόγραμμα βοήθειας θα μπορούσε να βοηθήσει και τους μικρούς γεωργούς ε, για να πολλούνται και τα δικά τους προϊόντα στα σχολεία, γιατί τα δικά τους προϊόντα είναι κατά κύριο λόγο τα πιο υγιεινά. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι αυτό ακριβώς ε, προβλέπει το πρόγραμμα. Δηλαδή υγιεινά, μη μεταποιημένα προϊόντα να προσφέρονται, να διατίθενται στα σχολεία. Ε, αυτά ακριβώς, σε αυτά που βλέπει αυτό το πρόγραμμα, ε, το εκπαιδευτικό και διατροφικό. Ο κύριος Ντόρμαν για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, υπάρχουν ε, πάρα πολλοί νέοι οι οποίοι ε, δεν την χάνουν ε, καλής και σωστής διατροφής ούτε και καταναλώνουν καλά τρόφιμα γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να στηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς τα παιδιά αυτά με τρόφιμα και μεγάλα το θέμα είναι ότι δυστυχώς δεν διαδίδονται πολύ αυτά τα προϊόντα. Επίση, ε, σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν ε, οικονομικά προβλήματα και γι' αυτό είναι δύσκολο ε, να πολλούνται αυτά τα προϊόντα. Βεβαίως πρέπει να διαφυλάξουμε τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας, αλλά οφείλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους νέους να ενημερωθούν το πώς χειριζόμαστε τα ζώα, η υγεία των ζώων είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Πρέπει να αποφεύγονται οι μεταφορές ζώων σε μεγάλες αποστάσεις. Πολύ ωραία. Ο κύριος Πίτερ Μαχ έχει το λόγο. Ένα λεπτό παρακαλώ. Αγαπητοί συναδελφοί, η πρόταση επιδότησης του γάλακτος για τα σχολεία είναι μια πρόταση που δεν μου αρέσει. Ε, νομίζετε ότι είστε σωτήρες των παιδιών και καφιέστε ότι δημιουργήσατε αυτό το εξαιρετικό πρόγραμμα, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μάνα μας που θα πρέπει να μας υπαγορεύει τι θα πρέπει να ε, τρώνε και να πίνουν τα παιδιά μας. Τα ωφέλη για την υγεία του γάλακτος είναι αμφισβητήσιμα και αν ε, πραγματικά θέλετε να δίνετε στα παιδιά ε, γάλα με γεύσεις δεν θα πίνουν μετά απλό γάλα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει τα χρήματα να μείνουν στις τσέπες των φορολογουμένων και να τα έχουν οι γονείς των παιδιών αυτών και να μην ανακατεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την περίπτωση αν ε, θεωρείτε ότι ε, πρέπει να γίνεται αυτό για τη χώρα σας, να το κάνετε σε εθνικό επίπεδο. Αν όμως ε, λέτε ότι πρόκειται για εθελοντικό πρόγραμμα, τότε οι χώρες που δεν θα συμμετέχουν έμεσα θα επιδοτήσουν τις χώρες που θα συμμετέχουν. Δέχεστε μια μπλε κάρτα, κύριε Μάντς, από τον κύριο Πόλτσεκ, το συμπατριώτη σας. Παρακαλώ κύριε Πόλτσεκ. Ευχαριστώ πολύ που δέχεστε και την γαλάζια κάρτα. Συνάδελφε, προσέξτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απαγορεύει τίποτα, απλώς ε, υποστηρίζει κάποια προϊόντα και νομίζω ότι αυτά θα ε, πρέπει να τα εξετάσουμε στο πλαίσιο των όσων μας είπατε. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αν υπάρχει ένα πρόγραμμα όπου διατίθενται 250 εκατομμύρια ευρώ για την επιδότηση συγκεκριμένων προϊόντων και τα προϊόντα αυτά θα περιλαμβάνουν και το γάλα ε, και θα υποχρεώσουμε τα παιδιά να πίνουν γάλα ε, εις βάρος άλλων τροφίμων και εις βάρος των φορολογωμένων που θέλουν να τους προσφέρουν κάτι άλλο. Ε, εντάξει, δεν απαγορεύουμε το σοκολατούχο γάλα, αλλά επιδοτούμε το γάλα το οποίο δεν θα το πίνει και κανές. Δέχεστε μία ακόμα μπλε κάρτα, κύριε Μάχ. Eh, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά που είπατε, συνάδελφε, και θεωρώ ότι είναι πονίδεστο το γεγονός ότι ένα τόσο καταπληκτικό πρόγραμμα ε, υποβιβάζεται κατά αυτόν τον τρόπο από εσά. Φαίνεται ότι είστε κάποιοι από τους λίγους εδώ που επικρίνουν το πρόγραμμα αυτό. Εγώ έχω παιδιά στο σχολείο και πραγματικά θα ήθελα όλα τα σχολεία να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό. Σας υπόσχομαι, κύριε ε, συνάδελφε, ότι ένα μήλο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα. Σας παρακαλώ λοιπόν, σταματήστε να να τη διαδικασία. Υποστηρίξτε το πρόγραμμα αυτό στα σχολεία και κάντε ό,τι μπορείτε για να προωθήσετε τον τομέα των απορροκυπευτικών και των φρούτων με ό,τι μέσο διαθέτεται. Αγαπητοί συνάδελφε, δεν καταλαβαίνω. Αν νομίζετε ότι τα μήλα και το γάλα είναι τόσο καλά για τα παιδιά σα, γιατί δεν του τα αγοράζετε να του τα δίνετε μόνοι σα. Γιατί πρέπει να επινοήσετε ένα πρόγραμμα για τα 500 εκατομμύρια ανθρώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρετε μήλα. Βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις. Ε, ζητάνε πολλοί συνάδελφοι μπλε κάρτα. Νομίζω ότι κανονικά θα έπρεπε να δίνει τη δυνατότητα για μία μπλε κάρτα σε κάθε ομιλητή για να διευκολύνουμε και τη συζήτηση. Ο κύριος Μάτο για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η συμφωνία αυτή είναι πολύ σημαντική για όλη την Ευρώπη. Είναι ένα πρόγραμμα ε, που επιδιώκει καλές διατροφικές συνήθειες. Πολύ καλό λοιπόν. πολύ δε περισσότερο που έχει αυξημένο προπολογισμό. Όμως υπάρχει κάτι άλλο έχει ιδιαίτερη σημασία για τι ε, ε, περιοχές, όπως τα κανένα νησιά από τα οποία προέρχομαι, γιατί αναγνωρίζει πως χρειάζονται περισσότερα κονδύλια για αυτές τις περιοχές, τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Για πρώτη φορά, στο πλαίσιο του ΠΟΣΕΙ, προβλέπεται ε, ένα κονδύλι για αυτά τα προϊόντα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βοηθούν περισσότερο αυτές τις περιοχές ε, για να τα, τις βοηθήσουν ε, δεδομένης της κατάστασής τους και της γεωγραφικής τους θέσης. Ε, εκεί η μεταφορά προϊόντων είναι πιο ακριβή, οπότε θα πρέπει να βοηθηθούν. ένα, επίσης είναι πολύ καλό για τους παραγωγούς μπανάνας. <laughs> Κάποιος είπε και με εξέπληξε ότι θα έπρεπε να διαγράψουμε την μπανάνα από τον τίτλο γιατί δεν παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, ασφαλώ και παράγεται. Παράγονται μπανάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τα Κανάρια νησιά παράγουν τι πιο νόστιμες μπανάνε του κόσμου και η Μαδέρα και η Μαρτινίκα. Μην τα ξεχνάτε αυτά. Θα σας φέρω μπανάνες από τα Κανάρια νησιά στην επόμενη ολομέλεια για να τις δοκιμάσετε, να τις δοκιμάσουν και αυτοί που αγνοούν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει μπανάνες. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια. Είναι πολύ σημαντικό που έγιναν αντιληπτές ιδιαίτερε ανάγκες των εξόχω απόκεντρων περιοχών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Περιμένουμε τις μπανάνες την επόμενη φορά. Ε, η κυρία Κιλέρα Γκαρσία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ε, συγχαρώ και εγώ τους συναδέλφους, ιδιαίτερα τον εισηγητή, τον κύριο Ταραβέλα. Έκανε πολύ καλή δουλειά μαζί με τους ε, σκιώδεις εισηγητές. Ε, δυσκολευτήκαμε να πείσουμε το Συμβούλιο ότι είναι πολύ σημαντικό να λεφτεί υπόψη η θέση μας. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η ανάγκη που υπάρχει να βελτιώσουμε τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών στην Ευρώπη. Οι διατροφικές συνήθειες είναι πολύ σημαντικό να αποκτώνται νωρί. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει ό,τι μπορεί. Επίσης, βοηθούμε και την ευρωπαϊκή παραγωγή. Η διανομή νοπών προϊόντων, η οποία έχει προτεραιότητα, με ευχαριστεί ιδιαίτερα. Αν λείπει κάτι στη διατροφή των παιδιών είναι τα νοπά προϊόντα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό το κριτήριο να, ε, είναι, να λαμβάνει ιδιαίτερη έμφαση. Επίσης, τα κριτήρια διανομής του γάλακτος ε, δεν λαμβάνουν υπόψη ε, τον αριθμό των παιδιών όπως λαμβάνει υπόψη στα προεκβευτικά. Κρίμα, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Επίσης, θα ήθελα να είχε συμπεριληφθεί και το ελαιόλαδο. Το ξέρει ο κ. Σταραμπέλα. Εν πάση περιπτώσει. Ε, συμπεριλήφθη στις εκπαιδευτικές προτάσεις. Χαίρομαι. Νομίζω ότι θα ψηφιστεί με πλειοψηφία αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ την κυρία Αγγιλέρα Γκαρσία. Ο λόγος του κύριο Τσάνι, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Ταραμπέλα. Ηράκλειος Άθλος. Σας ευχαριστώ πολύ και σας κύριε Ταραμπέλα και τους κοιόδης ηγητές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ασχοληθεί με τη διατροφή των παιδιών. Δεν γίνεται αλλιώς. Μιλούμε για 60 εκατομμύρια νέους και παιδιά στην Ευρώπη που δυστυχώς θα πρέπει να βοηθηθούν στην απόκτηση καλών ε, διατροφικών πρακτικών. Και είναι πραγματικά κρίμα που τα κράτη-μέλη δεν κάνουν ό,τι θα έπρεπε. Αν δεν είχαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, φοβάμαι ότι πολλά κράτη-μέλη θα είχαν απαλείψει, εξαλείψει τελείως αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ένα ακόμα σχόλιο. Ορισμένες χώρες ε, επιβάλλουν ΦΠΑ, για παράδειγμα 27% ΦΠΑ ε, στη χώρα μου, την Ουγγαρία, ε, σε αυτές τις διανομές, σε αυτά τα προϊόντα. Ας το σκεφτούμε. Θα πρέπει αυτού του είδους τα προϊόντα να μην υπόκεινται σε φορολόγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας το σκεφτούμε. Ε, Σας ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Σάνι. Και τώρα λοιπόν περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Μικολάσικ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. κύριε και κύριοι, εγώ πιστεύω ότι αυτό το πρόγραμμα για τα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ καλό. 1,5 δις ευρώ για 6 χρόνια, αυτό είναι το πρόγραμμα και αφορά 3 εκατομμύρια παιδιά. Δύο φορές την εβδομάδα θα παίρνουν ε, φρούτα, μπανάνες ή ε, γάλα και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους ε, νέους στην Ευρώπη. Όχι μόνο στις Ηνωμένε Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη τα παιδιά υποφέρουν από παχυσαρκία και αργότερα αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολλά προβλήματα υγείας. Ε, μπορεί να οδηγήσει σε κυκλοφορικά προβλήματα. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα ε, μπορεί εν μέρη να αναστείλει τέτοιου είδου προβλήματα. Χαίρομαι πάρα πολύ που το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν ε, θέσπισαν αυτή τη συμφωνία και το μέλλον πλέον είναι αισιόδοξο. Οι υγιείς, υγιεινές διατροφικές συνθήκες ενισχύονται, τα παιδιά θα αποφεύγουν τη ζάχαρη και θα ε, διατρέφονται πιο γίνα. Πολύ ωραία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τεραμπέλα για το πάθος του και για την επιμονή του γιατί με τον τρόπο αυτό μπόρεσε να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις. 250 ε, εκατομμύρια ευρώ, αυτό είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον και για την ανάπτυξη της κοινωνίας μας. Ε, η παροχή φρούτων και γάλακτος στα σχολεία αφορούν στην υγεία των παιδιών μας, τα οποία πρέπει να έχουν ισορροπημένη συγκεκριμένη διατροφή, να έχουν ε, ε, τρόφιμα με θρεπτική αξία και το σχολείο εδώ παίζει σημαντικό ρόλο. Ε, σήμερα με την παγκοσμιοποίηση η προσφορά είναι πολύ μεγάλη, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να εκπαιδεύουμε ενημερωμένους καταναλωτές για να αποφεύγουμε τις ασθένειες. Ευχαριστώ τον εισηγητή γιατί στον κανονισμό προτείνει και κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, δηλαδή τα προϊόντα που διανέμονται σχολεία θα πρέπει να είναι τοπικά από τοπικούς παραγωγούς για να ε, στηρίξουμε τους ε, γεωργούς, τους τοπικούς γεωργούς που έχουν υποφέρει πάρα πολύ και γιατί επίσης θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό οι ε, κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξοικειωθούν με τις παραδοχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Δείτε λίγο τι γίνεται με τις σκανδιναβικές χώρες. Τις χώρες μας ε, τα παιδιά μας ε, παίρνουν, λαμβάνουν υγιεινά σχολικά γεύματα τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω φορολογίας που σημαίνει ότι ακόμα και οι φτωχότεροι ε, της κοινωνίας μπορούν να απολεμβάνουν τέτοια σχολικά γεύματα για τα παιδιά τους. Το καλύτερο στο όλο σύστημα είναι ότι τελικά είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Εάν ένα παιδί ε, αποκτήσει υγιεινές διατροφικές συνέπειες και τις συνήθειες και τις ακολουθήσει αυτό στο μέλλον, τότε τα αποτελέσματα είναι σαφή. Λιγότερη παχυσαρκία, λιγότερες ασθένειες ε, και ε, λιγότερη επιβάρυνση και της οικονομίας τελικά. Νομίζω ότι αυτό τα οποία συζητάμε σήμερα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση πρέπει να υποστηρίξουμε τα υγιεινά τρόφιμα και τα υγιεινά γεύματα στα σχολεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ιβανίκοφσης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία στην ε, έκθεση αυτή. Ο κύριος Γιάκοφτσιτς και νομίζω ότι ήταν όλα πάρα πολύ ε, επιτυχημένα τα όσα προτίθηκαν και θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντική είναι η συγκεκριμένη έκθεση για να εκπαιδεύσουμε τους νέους μας ε, σε υγιεινές συνήθειες. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά τα οποία είναι σημαντικά για τους νέους μας. Επίσης ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω διότι αναγνωρίστηκαν και οι ανάγκες της Κροατίας και τα παιδιά στην Κροατία θα λαμβάνουν και αυτά επιτέλους αυτά τα οποία χρειάζονται. Υπάρχει όμως ένα στοιχείο το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό παρόλα αυτά. Το γεγονός ότι τα τοπικά ε, περιφερειακά προϊόντα θα διανέμονται στα σχολεία. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί πραγματικά ιδιαιτερότητα για τους νέους ανθρώπους, διότι θα μπορούν να αναγνωρίσουν που ζουν μέσω των προϊόντων τα οποία ε, χρησιμοποιούνται και παράγονται σε τοπικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Βιέγας. Είναι θετική η ιδέα από αυτό το πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά, η εφαρμογή του μπορεί να κάνει τη διαφορά. Δεν καταλαβαίνουμε ε, γιατί ε, τα δύο προγράμματα ενώθηκαν σε ένα. Οι, οι ζητούσαν δύο διαφορετικά προγράμματα. Δεύτερον, υπογραμμίζουμε ότι το πρόγραμμα αυτό θα πετύχει μόνο αν συνοδευτεί από μια ε, στρατηγική προς τοπικής ανάπτυξης, ε, τοπικών προϊόντων, κοινωνικής ε, και δαφικής ε, συνοχής στις τοπικές κοινωνίες. Η στρατηγική αυτή θα αποτύχει αν συνεχίσουμε να δεχόμαστε να υπάρχουν fast food έξω από τα σχολεία ή και μέσα στα σχολεία μηχανήματα τα οποία διανέμουν προϊόντα τα οποία πραγματικά δεν ε, είναι υγιεινά για τα παιδιά. Θα πρέπει να δώσουμε αυτό τον αγώνα για προς των παιδιών μας. Ευχαριστώ. Ε, Κυρία Ε, υποστηρίζω την ε, παροχή προεκπαιδευτικών γαλακτοκομικών και μπανανών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και συγχαίρω τον εισηγητή. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλε τι ευκαιρίε που μα δίδονται για να δίνουμε υγιεί εναλλακτικέ ε, στα παιδιά μα σε ό,τι αφορά τη διατροφή του. Με υγιεινέ ε, τροφέ για να καταπολεμήσουμε την παχυσαρκία. Όπω είπε και ο εισηγητή, βέβαια, τέτοιου είδου προγράμματα ε, δίδουν και δυνατότητα ε, εμπορία σε προϊόντων τα οποία αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στην εμπορία τους. Ε, είναι πολύ σημαντικό όμως να αυξήσουμε την συνειδητοποίηση ότι είναι καλά τα, και τα γαλακτοκομικά προϊόντα και όχι μόνο τα οπωροκυπευτικά. Ευχαριστώ. κυρία Σόιτροβα. Πρόεδρε, συμφωνώ με τους ε, προηγούμενους ομιλητές που ε, μίλησαν θετικά για το πρόγραμμα αυτό και για την έκθεση. Βλέπω ότι η έκθεση αυτή έχει την υποστήριξη σχεδόν όλων των πολιτικών ομάδων. Ε, το γεγονός ότι τα δύο προγράμματα συνενώθηκαν ε, δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς κονδυλίων και αυτό είναι πολύ καλό. Επίσης ε, διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογή ο αριθμό των προϊόντων τα οποία μπορούν να διανεμηθούν και συμπεριλαμβάνονται και μεταποιημένα φρούτα πλέον. Ο βασικός όμως και πρωταρχικός στόχος είναι η εκπαίδευση των ε, παιδιών ηλικιών από 6 έως 10 ετών. Να τα εκπαιδεύσουμε να, να τρώνε υγιεινές τροφές. πολύ συχνά οι γονείς ε, δεν έχουν τη δυνατότητα να δίνουν αυτά, να δίνουν αυτά τέτοιου είδους τρόφιμα, τροφές στα παιδιά. Οπότε πιστεύω ότι αυτό το πρόγραμμα θα βοηθήσει να βελτιώσουμε την υγεία των ε, παιδιών και βέβαια να προστατεύσει τα τοπικά προϊόντα. Ε, Ο κ. Νίκολα Καπούτο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ταραμπέλα για όλα αυτά που πέτυχε στο σημαντικό αυτό θέμα, δηλαδή την διανομή φρούτων και γάλακτος στα σχολεία. Ένα σημαντικό στοιχείο ε, που εξηγεί ότι έχουν πέσει, έχει πέσει η κατανάλωση αυτών των προϊόντων είναι ότι δεν τα διδάσκουμε στα παιδιά μας, δεν τους τα δίνουμε. Και αυτό συμπίπτει και με το ότι έχει αυξηθεί η παχυσαρκία διότι δεν καταναλώνουν προϊόντα που να είναι υγιεινά αλλά καταναλώνουν εκείνα που έχουν πολύ ζάχαρη. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να συγχαρώ ε, για όλα αυτά τα οποία αποφασίστηκα. Είναι πολύ σημαντικό να πλησιάσουν, να μάθουν τα παιδιά να πλησιάσουν τη γεωργία, να εξοικειωθούν και με την προέλευση προέλευση των προϊόντων, να εξοικειωθούν με τη γεύση ε, και με διάφορα προϊόντα, κυρίως ε, με τα προϊόντα της ε, περιοχής τους. Πρέπει να εξοικειωθούν και με τη διατροφική αξία. Εξάλλου, αυτό είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα για να διαδώσουμε αυτά τα οποία επιθυμούμε. Είναι ένα πρόγραμμα όπου τα κράτη-μέλη θα μπορούν και να ελέγχουν το τι γίνεται με όλα αυτά τα προγράμματα και έτσι ώστε αν υπάρξει κάποιο θέμα να μπορούν να αλλάξουν μακροπρόθεσμα ε, τα προγράμματα όσοι εφαρμόζονται. Ο Μαριάς παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο υποσυτισμός στην Ελλάδα έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. Σύμφωνα με το Ερευνητικό Ίδρυμα Πρόληψης, 6 στους 10 Έλληνες μαθητές το 2013-2014 δεν είχαν πρόσβαση σε τροφή επαρκούς ποιότητας επιπλέον για τη σχολική χρονιά δύο χιλιάδες το 53% των οικογενειών των μαθητών αντιμετωπίζουν επισητιστική ανασφάλεια και το 21% ένα πλήττονται από πείνα. αυτό αποδεικνύει ότι οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις για παροχή οπωροκυπευτικών προϊόντων ακόμη και γαλακτοκομικών προϊόντων στα σχολεία της ελλάδας είναι ημίμετρα και δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση του υποσιτισμού των παιδιών στην ελλάδα η οποία πλέον Ελλάδα αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια ανθρωπιστική κρίση πρέπει να καταστεί σαφές προ κάθε κατεύθυνση ότι η εξάλληψη του υποσιτισμού στα σχολεία δεν μπορεί να περιμένει καθώ η υγεία των παιδιών τίθεται σε κίνδυνο. αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι να βγάλει η τρόικα τη θηλιά του χρέου από την ελλάδα να σταματήσει η μερκελική λιτότητα και η ασφιξία τη ελληνική οικονομία, εν ώψη μάλιστα τη κρίσιμη κατάσταση που προκαλεί στην ελλάδα το προσφυγικό ζήτημα. ευχαριστώ. Ε, θα πρέπει να συμφωνήσω πως είναι πολύ θετικό βήμα η προσπάθεια που γίνεται ώστε να ενσωματωθεί στη διατροφή των Ευρωπαίων ενηλίκων η κατανάλωση σε μεγαλύτερο βαθμό νοπών οποροκυπευτικών φρούτων και φρέσκου γάλακτος. Βέβαια, πολύ αμφιβάλλω πως τα συγκεκριμένα μέτρα από μόνα τους θα φέρουν κάποιο αποτέλεσμα αν δεν συνδυαστούν και με μια ταυτόχρονη εκμάθηση των ευεργετικών αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης διατροφής όχι μόνο από τα παιδιά αλλά και από τους γονείς τους και τους υπόλοιπους ενήλικες. βεβαίως θα ήθελα να παρατηρήσω πως με τις πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζει η ευρωπαϊκή ένωση αυτή η διατροφή θα είναι ίσως και η μοναδική στην οποία θα έχουν πρόσβαση ορισμένα ελληνόπουλα μιας και έχουμε τεράστια αύξηση της ανεργίας και πολλοί γονείς αδυνατούν να προσφέρουν έστω και τα απαραίτητα στα παιδιά τους από τη στιγμή που έχουν μηδενικό εισόδημα ταυτόχρονα κράτος πρόνοιας δεν υπάρχει να μεριμνήσει για αυτούς καθώς οι ελάχιστοι διαθέσιμοι πόροι κατευθύνονται κατά προτεραιότητα σήμερα για την κάλυψη των αναγκών των μεταναστών. σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Ταραμπέλα, τους και και τον Επίτροπο γιατί Επιτέλους αυτό το πρόγραμμα γκρίθηκε και ένα πολύ σημαντικό μέτρο ως ελέγχτη γιατί με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθούν οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών και θα βελτιωθεί και η υγεία τους. Και από την άλλη θα καταστεί δυνατό τα φρούτα και τα λαχανικά να συμπεριλαμβάνονται ε, στο πρόγραμμα των σχολείων και αργότερα και στις οικογένειες. 250 εκατομμύρια ευρώ ε, αυτό ε, σημαίνει για τη Σλοβενία 300.000 περισσότερα ευρώ από την πέρυσι στην Σλοβενία. Με τον τρόπο αυτό ε, θα διατίθενται περισσότερα τοπικά ε, προϊόντα στα σχολεία. Αυτό λοιπόν το μέτρο μας δίνει πλέον τη δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται ποιοτικά προϊόντα όπως είναι το μέλι και είμαι πεπισμένος ότι τα κράτη-μέλη θα εκμεταλλευτούν αυτό το πρόγραμμα. Ο κύριος Σάντος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή η απόκτηση υγιών διατροφικών συνθήκων προωθεί τη βελτίωση της υγείας ε, και αν μιλάμε για τους νέους σίγουρα θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο της ε, δημόσιας πολιτικής ε, υγείας. Η διανομή αυτών των προϊόντων στα σχολεία αποτελεί πραγματικά κρατική επένδυση. Έχει και διπλό στόχο άλλωστε. διανομή τοπικών προϊόντων που θα ευνοήσει την τοπική παραγωγή με και ιδιαίτερα θετική διάκριση για τις εξόχως απόκεντρες ε, περιοχές ε, για τις οποίες προβλέπονται επιπλέον κονδύλια. Αυτό το σύστημα μπορεί να, είναι, να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικό, ιδιαίτερα λέω τη στιγμή της κρίσης σε ιδιαίτερου τομείς όπως για παράδειγμα του γαλακτοκομικού για τις ε, αζόρες που επίσης παράγουν μπανάνα θα μπορούσαν επίσης να αποτελέσει μια πρόσθετη βοήθεια για την διανομή τοπικών προϊόντων και του γάλακτος. Ευχαριστώ. Ε, ε, Τόμασιτς, η υγιής διατροφή ε, στα νηπιαγωγεία και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι ιδιαίτερο σημαντικό κομμάτι της ε, πολιτικής δημοσίας υγείας. Τα παιδιά μεγαλώνουν πολύ γρήγορα και θα πρέπει να αποκτούν διατροφικές συνήθειες από νωρί. Κρίμα που δεν είμαστε εξίσου ευαισθητοποιημένοι για το πώς το AIDS επηρεάζει την οικονομία μας. Ασφαλώς και θα πρέπει να διευκολύνουμε τη διανομή τέτοιων προϊόντων σε σχολεία και ιδιαίτερα στι πιο μειονεκτικές περιοχέ, Αλλά θα ήθελα να ενθαρρύνω τα κράτη-μέλη να απλοποιήσουν το φορολογικό του σύστημα ε, έτσι ώστε να βοηθήσουν τις εταιρείε να μην χρειάζονται τέτοιου προγράμματα. Αν τα παιδιά δεν, ζου, δεν έχουν γονείς που να δουλεύουν και να βγάζουν χρήματα, είναι χαμένα. Οπότε τις επιχειρήσεις που δίνουν δουλειές και απασχόληση θα πρέπει να βοηθήσουμε. Μόνο σε μια τέτοια ανταγωνιστική οικονομία μπορούμε να έχουμε εγγύηση για το μέλλον των επόμενων γενιών. Now on behalf of the European Commission, uh, Commissioner Phil Hogan. Take please. Ο κύριος Hogan, Ευρωπαϊκή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που υποστήριξαν και μάλιστα γενναιόδωρα το πρόγραμμα. Ε, το πρόγραμμα ε, προέκυψε από την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και από την έκθεση του Ευρωδικαστηρίου που είχε επισημάνει κάποιες παραλήψεις σε δύο προηγούμενα προγράμματα. Τώρα λοιπόν, επειδή θα ενοποιηθούν τα προγράμματα, θα εξοικονομήσουμε χρήματα, ε, θα έχουμε πιο αποτελεσματικά προγράμματα και θα μπορούμε να διοχετεύουμε τα κονδύλια απευθείας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εξάλλου, παρότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες ε, την ε, παραγωγή υπάρχει και αυξημένη ζήτηση ε, γιατί εφαρμόζονται αυτά τα προγράμματα στα κράτη-μέλη. Είναι ένα προαιρετικό πρόγραμμα, απευθύνομαι στους κυρίους Μακ και Άγνιου. Ε, κοιτάξτε, υπάρχει προαιρετική συγχρηματοδότηση. Δεν είναι δεσμευτικό ή υποχρεωτικό να χρηματοδοτούν τα κράτη-μέλη. Αυτό το έχει επιλέξει νομίζω το Ηνωμένο Βασίλειο. Αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στα τοπικά προϊόντα έναντι των για να έχουν καλύτερη υγεία τα παιδιά. Ακριβώς αυτό θέλει να κάνει το πρόγραμμα και αυτό κάνει. Κύριε κύριε Φραντζιλίκα και Μάτεο ανέφεραν τα φρούτα και τα λαχανικά πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων. Ε, συμφωνώ λοιπόν να συμπεριλαμβάνονται οι μπανάνες σε αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα γιατί αυτό είναι σημαντικό για περιοχές όπως είναι οι Κανάριες ε, νήσι αλλά και όλες οι εξόχως απόκεντρες περιοχές. Έτσι μπορεί να ε, βελτιωθεί, να αυξηθεί η κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προ την κυρία Γκραπίνη να σα πω ότι ο στόχο είναι τα παιδιά ηλικία 6 μέχρι 10 ετών. Ε, αυτό το πρόγραμμα ε, θα βοηθήσει να επιτευχθεί ο στόχος που θέλει και εκείνη ε, σε τόσο μικρή ηλικία επειδή θα εξοικειωθούν τα παιδιά ε, αργότερα θα μπορούν να αποκτήσουν καλές ε, υγιεινές συνθήκες όσον αφορά την ε, τροφή που θα καταναλώνουν. Ε, θα αποφύγουν την παχυσαρκία. Κύριε Γιάρ, συμφωνώ μαζί σας με αυτά που είπατε σχετικά με τον εξορθολογισμό του προγράμματος και θέλω να σας πω ότι το 2023 το πρόγραμμα θα αναθεωρηθεί. Κύριε Αγνιού, γνωρίζω ότι χρησιμοποίησατε τη λέξη κοινικός, αλλά όπως ξέρετε η γεωργοί στην, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν χρειάζεται να ανησυχούν γιατί παίρνουν 2,3 δις ε, το χρόνο από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους ε, και ελπίζω να συνεχίσουν να παίρνουν και στο μέλλον. Δεν ξέρω πώς θα τα συνεχίσουν να παίρνουν από το Υπουργείο Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου. Τέλος πάντων, ευελιξία κατά την άποψή μου θα βοηθήσει στο να είναι το πρόγραμμα πιο επιτυχημένο. Και στην κυρία Κίλε θέλω να πω ότι και το ελαιόλαδο συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα. Θα βοηθήσει τη χώρα που γνωρίζει πάρα πολύ καλά και προς την γαλλική αντιπροσωπεία να σας πω ότι και γαλλικά προϊόντα μέλη συμπεριλαμβάνεται έτσι λοιπόν ε, θα ε, βελτιωθεί και εκεί η παραγωγή Θεωρώ ότι θα υπάρχει ευελιξία. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ και πάλι τον κύριο Ταραμπέλα και τους και για τη συνεργασία που είχαμε και εύχομαι το πρόγραμμα να επιτύχει. Όπως και όλα τα άλλα προγράμματα θα αναθεωρηθεί το 2023. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ και τώρα ο εισηγητής, ο κύριος Ταραμπέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχά θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι πράγματι σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φροντίσαμε η νομική βάση να είναι μια βάση που να επιτρέπει σαφή συναπόφαση και να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους σκιώδη συζητητέ που με υποστήριξαν και τελικά καταφέραμε να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Όσον αφορά το περιεχόμενο, πέντε παρατηρήσει. Θα ήθελα να απαντήσω σε πέντε συναδέλφου που αναφέρθηκαν στα θέματα αυτά. Καταρχά, θα ήθελα να σα πω ότι υπάρχουν κριτήρια τα οποία μα επιτρέπουν να έχουμε... Ε, ε, στόχους για κάθε κράτος μέλος. Αλλά ε, τα, από 6 έως 10 ετών ε, το επιλέξαμε εμείς, αλλά μπορούν τα κράτη-μέλη κάλλιστα να επιλέξουν από την βρεφική ηλικία, από τον βρεφονιπιακό σταθμό ή αργότερα περνώντας στο δημοτικό σχολείο κλπ. Ε, δεύτερον, κάποιοι αναφέρθηκαν στο σοκολατούχο γάλα. Ε, μερικά γραμμάρια σοκολάτα σε κάτι πια δεν είναι τόσο βάνευσο Επίση, έχουμε επιμείνει να είναι πραγματική σοκολάτα, όχι χρωστική. Επομένω, αν με το σοκολατούχο γάλα τα παιδιά μπορέσουν να, να προσλάβουν περισσότερο ασβέστιο που κάνει καλό στην υγεία του, είναι καλύτερο. Τρίτον, κάποιοι επέκριναν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπαν ότι το Κοινοβούλιο εδώ ε, ακούει καλύτερα του πολίτε. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι όσον αφορά τη συγκεκριμένη πρόταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάστηκε πάρα πολύ καλά. Όπω και το θέμα του χειρού κρέατο που συζητάτε τώρα, ε, η Επιτροπή έκανε τη δουλειά τη, το Συμβούλιο είναι που καθυστερεί. Επίσης υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποιοι είπαν ότι η υγεία δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητα όταν σε 24 από τις 28 χώρες δεν υπάρχει κατάλληλη κατανόλωση φρούτων και λαχανικών καθημερινά και στα παιδιά αυξάνεται η παιδική πρεσυχησαρκία. Απλώς τους προτείνουμε λοιπόν και από εκεί και πέρα είναι ελεύθερα να επιλέξουν εθνική συγχρηματοδότηση. Πέμπτον, υπάρχει δυνατότητα συγχρηματοδότηση, όπω είπα και προηγουμένω. Ολοκληρώνοντα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τρία άτομα πιο συγκεκριμένα. Την Αλεξάνδρα Λεόνε, τη βοηθό μου, η οποία με βοήθησε πάρα πολύ, τη Μαρή Κουλτάρα από την πολιτική μου ομάδα και την κυρία Κουζινιέ από το ε, προσωπικό της Επιτροπής Γεωργίας ε, του Κοινοβουλίου που ήταν ιδιαίτερα δραστήρια κατά τη διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ταραμπέλα.